Muy buenos días. Comenzamos, se reanuda la sesión de la Comisión de, de Pesca. Con el punto de orden... Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με διάταξη παριθμό 14 την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Λαζάρου σε σχέση με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το κατά πόσο τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλαν στην προσαρμογή της ικανότητας των αλευτικών στόλων στις διαθέσιμες αλευτικές δυνατότητες. Η έκθεση αυτή είναι επικριτική όσον αφορά πολλές πτυχές της διαχείρισης. Παρίσταται εδώ ο κύριος ε, Λαζάρου για να παρουσιάσει την έκθεση και τις προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Ε, είχε προβλεφθεί και η παρουσία της κυρίας Επιτρόπου, της κυρίας Δαμανάκη, αλλά δεν μπόρεσε να παραστεί εδώ, γι' αυτό τροποποίησαμε την ημερήσια διάταξη. Ε, αλλά ε, δεν μπόρεσε να έρθει την Τετάρτη και μας παρακάλεσε να έρθει την ε, Πέμπτη. Και παρόλα αυτά, χθες το βράδυ μας είπε ότι δεν μπορούσε να έρθει χωρίς ε, να το δικαιολογήσει. Επίσης θα ήθελα να σε επενθυμίσω ότι η συνεδρίαση των συντονιστών του περασμένου Φεβρουαρίου αποφάσισε να γίνει μια έκθεση γνωμοδότησης για την ε, απαλλαγή ε, και ε, ανατέθηκε στον κύριο Μιλάνα από τους σοσιαλιστές. Θα έχουμε επίσης μια ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα για 40 45 λεπτά. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω καθυστερήσεις θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λαζάρου και προηγουμένως θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ. Thank you, Chairman. Uh, Chairman... Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αλίας. Πρώτα απ' όλα με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Φαίνεται ότι θα πρέπει να εξοικειωθούμε καλύτερα με, την, με το κυκλοφοριακό των Βρυξελών. Με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω την έκθεση 12 του ελεγκτικού συνεδρίου το 2011 με νέα μέτρα για να ε, προσαρμοστούν οι αλληλευτικές δυνατότητες στις διαθέσιμες αλληλευτικές ευκαιρίες των αλληλευτικών σκαφών. Η έκθεση αυτή έρχεται σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή για την κοινή αλληλευτική πολιτική εφόσον η πρόταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτής με το νέο Ταμείο της ε, Αλίας και της Θάλασσας είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβει υπόψη και η Επιτροπή σας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μπορεί να συνεισφέρει στις συζητήσεις σας η συγκεκριμένη έκθεση για αυτή την τόσο σημαντική μεταρρύθμιση. Εντάχει θα σας παρουσιάσω το ιστορικό της έκθεσης και θα ήθελα να τονίσω τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που κάνει το Ελληνικό συνέδριο. Ξεκινώντας με το ιστορικό. Επί σειρά ετών η τα αλληλευτικά αποθέματα και η αλληλεία ε, μειώνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλληλεία σε βιώσιμα επίπεδα έχει να κάνει και με την ε, μακροπρόθεσμη ε, βιωσιμότητα των αλληλευτικών πόρων και γενικότερα του αλληλευτικού τομέα. Με την πρόσφατη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής από το 2004 μειώθηκαν κατά ένα εκατομμύριο περίπου οι αλληλευτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάθηκαν 17.000 θέσεις εργασίας στον αλληλευτικό τομέα. Η υπερβολική δυνατότητα του αλλιευτικού στόλου έχει εντοπιστεί ως ε, ένας από τους βασικούς λόγους για την μείωση αυτή της ε, μετατροπής των ελευθερικών πόρων. Εδώ έγιναν πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, μεταξύ των οποίων η απόσυρση σκαφών και μέτρα περιοριστικά που επιβλήθηκαν στα κράτη-μέλη. Ωστόσο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ω τώρα δεν έχουν δώσει αποτελέσματα. Αυτό αναγνωρίζεται στην ε, πράσινη βίβλο τη Επιτροπή του Απριλίου 2009 με την ε, πρότασή τη για την τωρινή μεταρρύθμιση. Το ελεκτικό συνέδριο εντόπισε προβλήματα και με τι πλεονάζουσε δυνατότητε των στόλων ε, σε πρόσφατε εκθέσει του. Πιο πρόσφατα, μάλιστα, στην ειδική έκθεση υπαριθμών 7 του 2007 αλλά και από το 1993. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα που σήμερα κοιτάζουμε και εξετάζουμε ήδη υπήρχαν από πολλά χρόνια. Γνωρίζοντα ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική έπρεπε να μεταρρυθμιστεί ούτω ή άλλω και υπό το φω των γνωστών πλέον προβλημάτων, το Ελληνικό Συνέδριο αποφάσισε να μελετήσει νέα μέτρα για να ε, περιοριστεί η πλεονάζουσα δυνατότητα του ελληνικού στόλου ε, και την νομοθεσία τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Είδαμε τα ευρωπαϊκά μέτρα για να ε, προσαρμοστούν οι δυνατότητε του ελληνικού στόλου στι διαθέσιμε αλληλευτικέ ευκαιρίε. Τα 7 κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε, δηλαδή η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, από κοινού εκπροσωπούν περίπου το 70% των, ε, ε, της αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελευτικών δυνατοτήτων και 80% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Έτσι μας δίνουν μια πολύ καλή συνολική εικόνα για τις πλεονάζουσες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να περάσουμε τώρα στα βασικά συμπεράσματα. Το ελεγκτικό συνέδριο κατέληξε σε συμπεράσματα σε δύο βασικέ κατηγορίε. Πρώτον, σε σχέση με το πολιτικό πλαίσιο για τη μείωση τη πλεονάζουσα δυνατότητα του ελεκτικού στόλου. Και δεύτερον, σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων για να περιοριστεί αυτή η υπερβολική δυνατότητα. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Σε σχέση με το πολιτικό πλαίσιο. Πρώτον, δεν μετρήθηκε σωστά, δεν μετρήθηκαν σωστά οι δυνατότητε και οι πλεονάσει δυνατότητε του ελευτικού στόχου, στόλου. Ε, σε σχέση με, την, ε, με, την, ε, με τον όγκο και το μέγεθο. Εδώ δεν λήφθηκε υπόψη η αλλαγή των ελευτικών μεθόδων. Ενώ οι ονομαστικέ δυνατότητε των ελευτικών στόλων μειώνονται, η δυνατότητα του στόλου να αλλιεύσει τελικά αυξάνεται περίπου κατά 3% ετησίω. Αυτό εκτιμήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο ότι δίνει ένα αποτέλεσμα 60% αύξηση σε μια περίοδο 16 ετών, από το 1992 δηλαδή ως το 2008. Επιπλέον, την τελευταία φορά που μετρήθηκαν οι πλεονάσεις δυνατότητες του ελευτικού στόχου, πριν από 15 χρόνια, τότε υπολογίστηκε σε 40% με την τότε έκθεση. Αυτό ε, περιπλέκει το να γίνει σωστή στοχοθεσία για την μείωση. Ε, Επίση, τα ανώτατα όρια, προκειμένου να περιοριστεί το μέγεθο του ελεκτικού στόλου, ε, αρχίζουν να γίνονται άσκοπα. Έτσι λοιπόν τα ανώτατα όρια για τι δυνατότητες τις ενεργειακέ δυνατότητε και το μέγεθος του σκάφους είχαν τεθεί σε προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν είναι πλέον σκόπιμα καθώς ούτως ή άλλως το μέγεθος του στόλου είναι κάτω από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Θα έπρεπε Είμαστε ήδη σε 2.000 κυβικά μέτρα περισσότερο όγκο, αλλά παρόλα αυτά μένουμε εντό του πλαισίου. Έτσι λοιπόν ε, η κοινή ελευθερική πολιτική δεν έχει συγκεκριμένου κανόνε για το πώ αντιμετωπίζονται τα ελευθερικά δικαιώματα όταν αποσύρονται τα ελευθερικά σκάφη με κρατική επιχορήγηση. Έτσι λοιπόν Δίνονται αντιφατικά μηνύματα για το θέμα αυτό από την κοινή ελληνική πολιτική. Ο βασικό κανονισμό του Συμβουλίου από το 2002 προβλέπει την απόσυρση ελληνικών δικαιωμάτων για τέτοια σκάφη, όμω οι επόμενοι κανονισμοί που ορίζουν τι αιτήσει ποσοστώσει επιτρέπουν την επανακατανομή των δικαιωμάτων αυτών σε κάποιε περιπτώσει. κρατημέλη επιτρέπουν στου αλληλεί να πωλήσουν τα ελληνικά του δικαιώματα, ενώ άλλα τα απαγορεύουν η πώληση των αλληλευτικών ε, δικαιωμάτων των αποσυμμένων σκαφών ε, επιτρέπουν στους αλληλείς κάποιες φορές να, αναδιαρθρώσουν διαρθρώσουν τις ε, αλληλευτικές δραστηριότητες που τους απομένουν ή να επιδιώξουν άλλες δραστηριότητες βιοποριστικές. Όμως ο κανονισμός της κοινής ελευτικής πολιτικής δεν μας λέει τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αυτή όταν υπάρχει και κρατική βοήθεια για την απόσταση των σκαφών. επί της ουσίας, ο ρόλο των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών δικαιωμάτων στην περίπτωση τη χλωνέσια δυνατότητα του αλληλευτικού στόλου δεν διευκρινίζεται από την αλληλευτική πολιτική και τον κανονισμό τη. Στην εισαγωγή τη εκθεσή μα αναφερόμαστε στον κίνδυνο τη υπεραλίευση, κάτι που έχει να κάνει και με τα δικαιώματα ε, ε, πρόσβαση, τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί σωστά. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σημειώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν προσαρμοστεί σωστά οι ελευθερικέ δυνατότητε χωρί την χρήση κρατική βοήθεια και μέσω των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών δικαιωμάτων. Ε, μεταξύ των συμπερασμάτων μα, θεωρούμε ότι τα αλληλευτικά δικαιώματα είναι ένα θέμα που και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, ώστε να αντλήσουμε διδάγματα και από το παρελθόν. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφέρω μια ενδιαφέρουσα μελέτη που έχει ετοιμαστεί για το ε, Κοινοβούλιο, τίτλο 2. Ε, για την διαχείριση της αλίας και η οποία εντοπίζει παρόμοιε συστάσει με τη δική μα έκθεση. Υπάρχουν κάποια σημεία τώρα τα οποία θα ήθελα να τονίσω με συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί πλεονάσια δυνατότητα του αλληλευτικού στόλου. Πρώτον, υπήρξαν καθυστερήσει στην υλοποίηση και την εκτέλεση των κομπηλίων ε, του Κοινού Ελευτικού Ταμείου ε, από τα κράτη-μέλη. Ε, μέχρι το 2008 μόνο 645 εκατομμύρια από το διαθέσιμο ποσό του ενός δις περίπου ευρώ ε, αξιοποιήθηκαν επιπλέον τα κράτη-μέλη με τα λειτουργικά τους προγράμματα και τους στόχους που πρέπει αυτά για τη μείωση των στόχων δεν δικαιολόγησαν επαρκώς παραπέμποντας στην ε, κατάσταση των ελευτικών πόρων. Επίσης υπήρξαν προβλήματα με τις ε, προγράμματα προσαρμογής των ελευτικών προσπαθειών με συγκεκριμένους μηχανισμούς για την διαχείριση των ελευτικών σκαφών για παράδειγμα ορίστηκαν ε, στόχοι μείωση τη ελάχιστη δυνατότητα των σκαφών ε, που δεν έγιναν πάντα τότε σεβαστοί. Το βασικό ε, θέμα εδώ είναι ότι δεν υπήρξε επαρκή σχεδιασμό για τα λιευτικά σκάφη από την πλευρά τη Επιτροπή και με κρατική βοήθεια. Τα μέτρα δεν ήταν επαρκή. Third. Τρίτον, οι επενδύσεις επί των σκαφών για την αύξηση των ε, ε, αλληλευτικών δυνατοτήτων των σκαφών δεν είναι επιλέξιμα για κρατική βοήθεια. Τελικά χρηματοδοτούνται κάποιες φορές. Όπως με τη χρηματοδότηση καλύτερων ε, συστημάτων που επιτρέπουν στα σκάφη να αλλιεύουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα από ό,τι στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, εφόσον η κρατική βοήθεια αξιοποιείται για την βελτίωση τη ελευθερική δυνατότητα, αυτό αντιφάσκει με, του στόχου περιορισμού των ελευθερικών δυνατοτήτων. Επιπλέον, το μητρό των ελευθερικών σκαφών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το νεολόγιο, δεν έχει ενημερωθεί σωστά σε σχέση με του στόχου απόσυρση σκαφών. Και τα ανώτατα όρια δεν έγιναν πάντοτε σεβαστά. Έπειτα, ε, πέμπτο, ε, ενώ μεταξύ του 2003 ε, και του 2009 5.800 σκάφια αποσύρθηκαν, ε, μάλλον λειτουργούσαν με μεγάλη δυνατότητα χωρητικότητας, ε, τελικά ενώ ήταν επιλέξιμα για απόσυρση αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν είχε όμως μεγάλο αντίκτυπο στους αλλιευτικούς πόρους. Σε κάποιε φορέ, μάλιστα, δόθηκε κρατική βοήθεια για αλλιευτικά σκάφη, τα οποία ήταν ήδη αδρανή και Υπήρξαν σκάφη τα οποία αλλιεύαν ε, ε, αμεληταία ποσοστά των αλλιευτικών πόρων που είχαν εντοπιστεί. Εδώ κρατική βοήθεια δόθηκε με ένα από τα κράτη-μέλη και αυτό εντοπίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στι νέε προτάσει για το Ταμείο Αλία και Θάλασσα η Επιτροπή ε, αποφάσισε ότι η αντιμετώπιση τη της κρατική βοήθεια και των πλεονάζουσων δυνατοτήτων για να Ε, μείωση τη πλεονάζουσα δυνατότητα οδήγησε στην σπατάλη 1,7 δι ευρώ. Επίση, η ελοποίηση του κανονισμού ε, οδήγησε σε ανεπαρκή αποτελέσματα, διότι θα μπορούσε να δίνει μεγαλύτερα κονδύλια για τον εξυγχρονισμό των σκαφών και την απόσυρσή του, αλλά τελικά το 2008 πολλές φορές ε, επιβαρύνθηκε και από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Το ελεκτικό συνέδριο εντόπισε ότι οι όροι και οι δυνατότητες δεν οδήγησαν σε των μέτρων αυτών δεν οδήγησαν στη σωστή, στο σωστό περιορισμό των πλεονάζουσων δυνατοτήπων με την ε, επιλογή ακατάλληλων σκαθών. Επίσης, οι κανόνες για τα κράτη-μέλη και, τους, και τα μέτρα που προβλέπονται για την μείωση της, ε, των δυνατοτήτων υπεραλίευσης των κρατών μελών είναι ανεπαρκή. Οι εκθέσεις που προβάλλουν τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται πολλές φορές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν αδύνατο να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες για την υπεραλίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις εκθέσεις μας που τα τι συστήνει λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο. Η έκθεση συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί πολύ σοβαρά εάν πρωτοβολίε ή αναθεωρήσει των βασικών κανονισμών απαιτούνται και να ορίσει καλύτερα τα μέτρα για την αντιμετώπιση τη υπεραλίευση και των πλανοδοσών ελεκτικών δυνατοτήτων. Να λάβει μέτρα για να αναχαιτήσει την υπεραλίευση, να, να ορίσει πραγματικά όρια ρεαλιστικά για την περιορισμό των ελευτικών δυνατοτήτων των ελευτικών σκαφών, να ξαναδεί τα δικαιώματα μεταβίβασης ε, αλλήλευση και επίσης τον εξυγχρονισμό των σκαφών. Ακόμη να βελτιώσει την ποιότητα των μητρώων των ελευτικών στόλων και τις προσπάθειες για την εξωσορρόπηση των ελευτικών δυνατοτήτων που πλεονάζουν με αλληλευτικές ευκαιρίε. Η έκθεση καταγράφεται τα κράτη-μέλη υλοποιούν εγκαίρο, θα πρέπει να ε, υλοποιούν εγκαίρω τα μέτρα του αλληλευτικού ταμείου και οποιαδήποτε χρηματοδότηση και στήριξη, βελτίωση μάλλον των αλληλευτικών δυνατοτήτων των σκάφων δεν θα πρέπει να αυξάνεται την αλληλευτική του δυνατότητα. Θα πρέπει καλύτερα να εφαρμόζουν τα προγράμματα των, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ε, καταφέρουν να περιορίσουν τις πλεονάζουσες δυνατότητες. Εδώ πιστεύουμε ότι δεν θα πετύχουν τα μέτρα αυτά της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πλεονάζουσας δυνατότητας αλληλεύσης. Εδώ πρέπει να εντοπιστεί σε τι βαθμό υπάρχει η δυνατότητα αυτή, το ποσοστό υπεραλίευση, να ληφθούν ρεαλιστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί και να καταγραφούν σωστά οι επιδόσει. Η σημερινή μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική, τη κοινή αγροτική ε, πολιτική όπω προτείνεται και οι σχετικέ διευθετήσει ε, λαμβάνει υπόψη και το πρόβλημα τη υπεραλίευση και ελπίζουμε η έκθεση αυτή να συνεισφέρει στην όλη διαδικασία. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσει. Ευχαριστούμε, πολύ κύριε Λαζάρο. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω στο λόγο στον κύριο Μιλάνα που είναι ο εισηγητής αυτής της ε, έκθεσης. Ο κύριος ε, Μιλάνα δεν ε, παρίσταται όμως μου έδωσε την παρέμβασή του την οποία θα συνοψίσω εγώ, θα σας παρουσιάσω συνοπτικά. μιλώ λοιπόν εξ ονόματος του κυρίου Μιλάνα. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, εξετάζει κατά πόσο η προσπάθεια της ε, Επιτροπής στο πλαίσιο του προγραμματισμού ε, των κονδυλίων μπόρεσε να μειώσει την υπεραλίευση. Η μείωση της αλληλευτικής ικανότητας σε όγκο και σε ισχύ των κινητήρων αντισταθμίστηκε από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θεωρεί ότι η μείωση που έχει σαν στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον όγκο ήταν 29% το 2008, ενώ η αύξηση της πραγματικής αλευτικής ικανότητας ήταν 43% στην ίδια περίοδο, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτή η αύξηση είναι υπεύθυνη για μια εξοικονόμηση τάξη του 14% των πόρων. Λόγω του εξοχρονισμού του στόλου με τα κοινοτικά κονδύλια αυξήθηκε η αλευτική ικανότητα, αλευτική ικανότητα των σκαφών και ε, πολλές φορές δεν υπήρξε σωστή επιλεξιμότητα των ε, στόχων. Ο ευρωπαϊκός ε, στόλος είναι υπέρ μεγέθης και βρισκόμαστε μακριά από το στόχο μιας βιώσιμης διατηρήσιμης αλίας. Θα πρέπει να μειωθεί η ελευτική ικανότητα, να προσαρμοστεί στις πραγματικές αλευτικές δυνατότητες των αεροσκαφών και, ε, των ε, ε, αλληλευτικών σκαφών και στην διατηρησιμότητα των αποθεμάτων. Θα πρέπει να καταβληθεί μια προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών στη βάση της πραγματικής αλληλευτικής ικανότητας και της επίπτωσης του σπόρου της ευρωπαϊκής κοινότητας. Θα πρέπει τα αλληλευτικά σκάφη να προσαρμοστούν ανάλογα και θα πρέπει να οριστεί η διαχείριση των αλληλευτικών δικαιωμάτων σε σχέση με τον αριθμό των αλληλευτικών σκαφών που έχουν αποσυρθεί με τα κονδύλια των ε, δημόσιων πόρων. Τα κονδύλια τα οποία θα λάβουν οι πλειοκτήτες ε, ε, θα γίνει μέσω του συστήματος ατομικά μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων. Υπάρχουν δύο τύποι ερωτημάτων. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν καταλαβαίνει γιατί ε, το θέμα αυτό ανατέθηκε στην ε, Επιτροπή χωρίς να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Αλίας. Δεν ε, προβλέπονται επίσης αντισταθμίσεις για τους αλείς σε περίπτωση παραπλησμού των σκαφών. Ε, δεύτερον, ε, στην ε, Μεσόγειο οι προϋποθέσεις αλίας δεν μπορούν να βασίζονται στις ποσοστώσεις αλιεύματος, αλλά θα πρέπει να συνδυαστούν με το, αλευτικό, με το Ταμείο Αλίας. ζητούμε να υπάρξει μια περίοδος μεταβατικής μείωσης των κονδυλίων σε σχέση με την απόσυρση των αλλιευτικών σκαφών. Η μείωση της αλλιευτικής ικανότητας είναι μόνο μία από τις παραμέτρους για μία πραγματική μείωση της υπεραλίευσης που έχει άμεση επίπτωση στη διατήρηση των αποθεμάτων. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουμε κάποια συμπληρωματικά μέτρα ούτε ώστε να μειωθεί ο στόλος και να προχωρήσουμε στην προσωρινή αναστολή των ε, αλευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες ε, ε, περιόδους, δίδοντας δημόσιες ενισχύσεις. Ε, επίσης, η αλία θα πρέπει να μειώνεται κατά τις φάσεις ε, αναπαραγωγής των ηχθείων. Θα πρέπει να υπάρξουν τοπικά προγράμματα διαχείρισης της αλίας και να υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα για την επιβίωση των αλίων, τουριστικές δραστηριότητες κλπ. Ε, θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η χρήση κάποιων πιο επιλεκτικών αλληλευτικών εργαλείων, πιο συμβατών με την ε, διατήρηση του περιβάλλοντος. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έλαβε ε, υπόψη του τις διάφορες μορφές αλλίες και τους διάφορους, τα διάφορα είδη χθείων. δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια μοναδική λύση όσον αφορά την υπεραλίευση ε, υπάρχει μια κατάσταση ολιγοπολίου σε σχέση με, την, το μειωμένο αριθμό των φορέων και δεν ενδείκνει τα μέτρα αυτά για την αλία μικρής κλίμακας. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν επικεντρώνεται ε, στο κόστος το οποίο συνεπάγεται η απόσυρση των σκαφών. Και λυπάται για το γεγονός ότι οι δείκτες της ελευτικής ικανότητας ε, σε σχέση με την αλία ανοιχτή θάλασσα σε συνάρτηση με την ισχύ των κινητήρων των ελευτικών σκαφών δεν έχει ληφθεί υπόψη και συνεπώς δεν έχει καταρτιστεί, εκπονηθεί ένα ενδεδειγμένο πρόγραμμα δράσης. Αυτή ήταν η παρέμβαση του κυρίου Μιλάνα και κλείνοντας θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές που μας ζήτησαν το λόγο. Έχουμε τέσσερα αιτήματα. Καταρχήν ο κύριος ε, Καντέκ. Κύριε... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαζάρου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, όπου και αν είναι, αναγνώσκεται με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να διαβάζει κανείς και ανάμεσα στις γραμμές. Πάντως καταλήγει σε διαπιστώσεις και σε συστάσεις. Μας λέτε ταυτόχρονα δύο πράγματα. Ότι η πλεονάζουσα χωρητικότητα δεν είναι ορισμένη και ταυτόχρονα λέτε ότι πρέπει να την μειώσουμε. Ε, τι εννοείτε. Μου φαίνεται παράξενο. Εξάλλου, από όσο γνωρίζω και εσείς κύριε Λαζάρου το είπατε, δεν είναι ακριβώς γνωστή η χωρητικότητα η αλληλευτική ικανότητα. Δεν λέω περισσότερα γιατί δεν είναι γνωστός ο ορισμός της. Άρα, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε στο τι είναι αυτή η πλεονάζουσα χωρητικότητα. Και τι σημαίνει για την βιωσιμότητα της αλίας που όλοι αυτό θέλουμε. Και πρέπει να είναι βέβαια προσαρμοσμένη και σε κάθε είδος αλίας. Αν τώρα πράγματι υπάρξουν περιπτώσεις πλεονάζουσας χωρητικότητας, οι λύσεις μας λέτε δεν είναι υποχρεωτικά ίδιες από ένα στόλο σε άλλο και από μια χώρα σε άλλη. Και οι μεταφερόμενες ε, αλληλευτικές παραχωρήσεις και αυτές δεν είναι απαραίτητα η λύση. Εγώ νομίζω ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει τα δικά της μέτρα για τον παροπλισμό των ε, σκαφών. Ο Γκουίντο Μιλάνα τα λέει επίσης στην εκθεσή του δεν έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, λέτε. Μα ναι, αν δεν είχαν υπάρξει τα σχέδια αυτά, δεν ξέρω πόσα πλοία, πόσα σκάφη θα είχαμε σήμερα. Είπατε για 70.000 ε, θέσεις εργασίας και 386 σκάφη. Εγώ νομίζω, δυστυχώς χτυπάνε τηλέφωνα και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Επίσης η αξιολόγηση, οι, οι επιχορηγήσεις για τον εξυγχρονισμό είναι αρκετά ασαφή αυτά. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουν αυτά και για λόγους ασφαλείας βέβαια, αλλά και για λόγους κατανάλωσης ενέργειας, εκπομπής καυσαερίων και άλλα. Είναι στοιχεία ενός εξυγχρονισμού, αν θέλουμε μια βιώσιμη αλία αλλά σύγχρονη ή καθόλου αλία. Υπενθυμίζω μόνο ότι στην έκθεσή σας δεν βλέπω πουθενά το γεγονό ότι ο συντάκτης καταλήγει στο ότι πρέπει να θεσπιστούν παραχωρήσεις, μεταφερόμενες παραχωρήσεις για την αλία. Και μπορώ να τα διαβάσω όλα, αλλά δεν βλέπω πουθενά για επιχορηγήσεις για τον εξυγχρονισμό. Και σε ορισμένα άρθρα μάλιστα λέει ότι τα σχέδια παροπλισμού έδειξαν την αποτελεσματικότητά τους, ιδίως για τους πελαγικούς τόλους. Πάλι με κάποια προσοχή αυτό, τα συμπεράσματα της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρέπει να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα και από τα συμπεράσματα αυτά σίγουρα θα προκύψουν, θα προκύψουν οι διατάξεις του βασικού κανονισμού για τη μελλοντική αλληλευτική πολιτική. Εγώ πάντως αυτά τα πράγματα βρίσκω να λείπουν από την έκθεση που διάβασα. Πάντως, κύριε Ζάρο, σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που δώσατε. Εσείς κύριε Στίβενσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Λαζάρου που ήρθε σήμερα εδώ να μας μιλήσει. Δύο ή τρία σχόλια. Είπατε στην αρχή της Παρουσιάσω σα ότι μειώθηκαν τα αλλιεύματα κατά ένα εκατομμύριο τόνους από το 2002 που έγινε η προηγούμενη. Η έστη ECF που μας δίνει τις επιστημονικές σύμβουλες βρίσκει 30% αύξηση των εμπορεύσιμων αλλιευμάτων. Εγώ είχα πάει προ στην Ολλανδία και επισκέφθηκα ένα λιμάνι, το ΕΡΚ, στο βόρειο μέρος της χώρας αυτής και οι ψαράδες μου είπαν ότι υπάρχει πιο πολύ χωματίδα στη Βόρεια Θάλασσα και πιο πολύ ρέγγα από ό,τι έχουν δει εδώ και πολλά χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι παλεύουν με τα πεπαλαιωμένα σκάφη, της στράτες τους τις παλιές και δεν έχουν λεφτά για να αντικαταστήσουν τα σκάφη αυτά και να συνεχίσουν την αλία. Μάλιστα, επινόησαν ένα νέο τρόπο αλίας για να ψαρεύουν την χωματίδα, αλλά δεν έχουν λεφτά για να ε, εξοπλίσουν τα σκάφη τους, γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν τα παλιά σκάφη, κανένας δεν τα θέλει. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να εξετάσουμε όντως το πρόβλημα της άουσας χωρητικότητας, αλλά Εκεί που είδα εγώ το πρόβλημα αυτό στο ΕΡΚ ή αφήνουμε την αγορά να τα ρυθμίσει ώστε οι άνθρωποι αυτοί πλέον θα χάσουν τα προστοζήν δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα σκάφη και αυτές οι παλιές στράτες δεν είναι οικονομικές πλέον και θα καταρρεύσει ολόκληρη αυτή η κοινότητα ενώ υπάρχει πολύ χωματίδα στη Βόρεια Θάλασσα. Πώς το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Γιατί αν απλώς βγούμε και πούμε το πρόβλημα είναι πλεονάζουσα χωρητικότητα και άρα αυτό το πρόβλημα πρέπει να λύσουμε και θα λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς με τις ε, μεταφερόμενες αλληλευτικές παραχωρήσεις θα ζημιώσετε κοινότητες όπως αυτές του ΕΡΚ. Επίσης, και εδώ αρχίζω και αντιμετωπίζω πρόβλημα με όλα αυτά, μου είπαν ότι λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων πρέπει να επενδύσουμε σε καλύτερες μηχανές για τα σκάφη αυτά, για να μειωθούν και οι καταναλώσεις, να, κατα... μειωθούν και οι αερίων του θερμοκηπίου. Εγώ έχω πάει σε πολλά λιμάνια στην Ευρώπη, ως εισηγητής της ΕΜΟ, και είδα σκάφη που λένε ότι έχουν 300 ύπους υποδύναμη, ενώ στην πραγματικότητα έχουν πόρτες των 100 κιλών που κρέμονται από τις πλευρές των σκαφών τους. Με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσαν να κινήσουν τέτοια σκάφη με οι μηχανές των 300 ύπων. Αν λοιπόν όντω μας ενδιαφέρει ο εξυγχρονισμό των μηχανών για να βελτιωθεί η κατανάλωση ενέργειας, ε, να μειωθούν οι ρήποι κτλ. Πρέπει να επιμείνουμε σε μια πραγματική μέτρηση των υποδυνάμεων. Δεν έχει νόημα να λένε ότι έχουν πολύ περιορισμένες υποδυνάμεις Προφανώς είναι ψευδεί οι δηλώσει αυτές. Έχουν πολύ μεγαλύτερε υποδυνάμεις τα σκάφη αυτά. Και το άλλο σημείο κριτικής ε, επί της εκθέσεώς σας, αν με επιτρέπετε, τα αποθέματα των ψαριών άρχισαν να μειώνονται από το 62 και πουθενά στην έκθεσή σας δεν είδα καμιά αναφορά στην κλιματική αλλαγή, στην ε, ρήπανση της ε, θάλασσας, στη μείωση της περιεκτικότητας ε, σε οξυγόνο, την όξυνση των θαλάσσιων νερών, την οξύνηση μάλλον. Έχουμε πολύ, πολλά στοιχεία συλλέξει στην Επιτροπή Αλίας εδώ και πολλά χρόνια για τη μετακίνηση των αποθεμάτων του γάδου από τη Βόρεια Θάλασσα που έφυγαν 200 μίλια πιο ψηλά γιατί έχει ζεσταθεί η Βόρεια Θάλασσα. Είναι υπερβολικά θερμά τα νερά της για αυτά τα ψάρια. Οι ψαράδες όλο και περισσότερο δυσαρεστούνται, απογοητεύονται, διότι όλο το βάρος των ευθυνών το ρίχνουμε πάνω τους. Αυτή υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνοι για την υπεραλίευση, άρα πρέπει να περιοριστεί η πλονάζουσα χωρητικότητα των σκαφών τους. πολύ κύριε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Λαζάρου, που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Ακούσαμε την περίληψη της έκθεσης και της συστάσεις, αλλά εδώ διαπιστώνω ότι αναφέρεται ένας αριθμός χωρών. Ε, Περίεργως η Ιρλανδία δεν συμπεριελήφθη, θα θέλαμε να είχαν μελετηθεί και οι δυνατότητες της Ιρλανδίας, να ξέρουμε πώς θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σωστά τα κριτήρια στο μέλλον. Η κατάσταση στην Ιρλανδία πραγματικά ε, ανταποκρινόταν σε πραγματικό ε, παροπλισμό. Υπήρξε παροπλισμό. Θα πρέπει βεβαίω να υπάρξει καλό σχεδιασμό και μελέτη, όπω είπατε, για τα μέτρα τη Επιτροπή. Αλλά τα μέτρα που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Μεσόγειο Θάλασσα, λόγου χάρη, δεν είχαν τα σωστά αποτελέσματα. Ακριβώ γιατί δεν υπήρξε σωστή στοχοθεσία. Σε εμά, στην Ιρλανδία, με την αρμόδια επιτροπή για την Αλία, υπήρξαν ε, τέτοιε μελέτε στοχοθεσία και ένα μέρο ήταν από τα ε, από θέματα που υπάρχει πίεση να αντιμετωπίσουμε εκεί ακριβώ την ε, πλεονάζουσα δυνατότητα του στόλου. Το 30% των ε, δυνατοτήτων ε, των ε, βαθυπελαγικών δυνατοτήτων μειώθηκε. Αυτό σημαίνει ότι οι ποσοστώσεις που αλλιεύονταν μοιράστηκαν στο υπόλοιπο 70%. Άρα υπήρξε περισσότερο κέρδος διότι έτσι εξισορροπήθηκε η ανάγκη της απώλειας. Σε μια πρώτη φάση υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση και μετά υπήρξε κέρδος. Η... Για τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα δεν είναι αυτή η λύση η Επιτροπή να εγκρίνει τους δύο κανονισμούς απλώς. Το θέμα δεν είναι να, γίνουν, να κάνουμε τους πλουσιότερους ε, ακόμη πιο πλούσιους και τους στοχούς είναι σφάλμα να πιστέψουμε ότι αν αγοράσουμε τα ατομικά μεταβιβάσιμα δικαιώματα κάποιων αυτών, αυτό θα λύσει το πρόβλημα γενικώ. Όχι, η χωρητικότητα σε τόνους πρέπει να ελέγχεται. Υπάρχει άμεσο συγχετισμό εδώ μεταξύ των ποσοστώσεων που τα αλλιευτικά σκάφη επιτρέπεται να αλλιεύουν και του ελέγχου που γίνεται. Είναι σαν να υποθέτουμε ότι τα σκάφη που έχουν μια συγκεκριμένη δυνατότητα μπορούν να αλλιεύουν ε, όσο θέλουν. Ό,τι αλλιευτικό απόθυμα του ζητήθηκε να το αλλιεύουν. Αλλά δεν είναι έτσι το σωστό, διότι τότε τα κράτη-μέλη θα έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό συνέβη, συνέβαινε κάποτε σε κάποιε χώρε, αλλά έχουν αλλάξει οι καιροί. Οι αλλιεί έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να αλλιεύουν ακριβώ μέσα στα όρια τη ποσότητα που του έχει αποδοθεί και που του επιτρέπεται. Και αυτό για να διατηρούνται σε σωστά επίπεδα οι τιμέ. Βεβαίω κάποιοι αλλιεύαν ε, λαθρέω και αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι τιμέ ε, των ε, των προϊόντων τελικά κατέληγαν και στα νόμιμα και στα μαύρα, στα παράνομα να μειώνονται. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία να το μελετήσουμε αυτό. Έχει εδώ ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω, αλλά και κάθε κάτω μέλο για τον έλεγχο με ικανοποίηση σημειώνω, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω εγώ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον το ελεκτικό συνέδριο δεν επενεί ιδιαίτερα τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα. Και αυτό που ερμηνεύω εγώ, για να πάω λίγο παραπέρα με τις συστάσεις είναι να μην σταματήσει η απόσταση, να μην σταματήσει ο παροπλισμός. Οπότε δεν μπορούμε να τρέξουμε στο ελεγκτικό συνέδριο και να πούμε ότι το είπατε κι εσείς ως επιχείρημα. Δεν το έχετε πει. Ναι, εγώ λέω να υπάρξει παροπλισμός ε, και, το, και επιμένω σε αυτό. Και στοχοθεσία. Στοχοθεσία συγκεκριμένα ήδη. Σταθερή, σαφή στόχη, εν, εν, εντατακοποίηση των προσπαθειών και τελικά θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Θα πρέπει φαντάζομαι ως ε, ελεγκτές να κοιτάζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Είναι μεγάλο το ζήτημα ε, που πρέπει να καλύψει τα βάσιμα τα δικαιώματα. Θα μπορούσαν ε, χώρε σαν τη δική μου να δώσουν όλες τις δυνατότητες και τελικά να προχωρήσουν. Αλλά έτσι θα αυξηθεί μόνο η ποσόστοση. Οι κάτοχοι των σκαφών, οι πλειοκτήτες, μπορεί να έχουν ένα μέσο, άμεσο, ένα βραχυπρόθεσμο εισόδημα έτσι, αν πουλήσουν τα δικαιώματά του. Αλλά τι θα κάνουν αυτοί που απασχολούν και τι θα κάνει η ελευθερική βιομηχανία γενικότερα, οι μικροί και οι μεσαίοι λιμένε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Όλε αυτέ ε, τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα θα πάνε σε μεγαλύτερε χώρε, σε μεγάλε εταιρείε και αυτοί που ζουν στι περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά θα χάσουν. Θα μείνουν απ' έξω. Ιδιαίτερη ικανοποίηση λοιπόν σημαίνω, δεν ταχθήκατε υπέρ των μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων και ελπίζω αυτό να το λάβουν υπόψη και η Ευρωπαϊκή, υπόψη και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη και το Συμβούλιο. Ε, στοχοθετημένη λοιπόν εδώ απόσυρση, παροπλισμός, διότι εδώ η στοχοθεσία είναι ο καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε την επίτευξη των στόχων μα, να αυξήσουμε τι ποσοστώσει για αλληλευτικά σκάφη που θα μείνουν ε, στην ε, όλη δραστηριότητα τη αλληλεία μετά τον παροπλισμό. Και ελπίζουμε ότι συνολικά θα υπάρξει θετική, θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι σας είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων για την έκθεση αυτή, γιατί θεωρώ ότι μας πέστε την προσοχή σε κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε εντοπίσει εμείς από μόνοι μας. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει βεβαίως τώρα να τα αξιολογήσουμε από πολιτική άποψη και ασφαλώς θα το πράξουμε. Θεωρώ ότι γίνεται πολύ ξεκάθαρο και στη δική σας έκθεση ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, που υφίστανται και στο παρελθόν ήταν ολέθριες και συνεπώς ε, είναι δικό μας επιτεκτικό μέλημα στο πλαίσιο της νέας μεταρρύθμισης να εκπονήσουμε νέα εργαλεία για να μειώσουμε την υπεραλίευση. Και σας είμαι ευγνώμων που μας λέτε ότι θα πρέπει να ορίσουμε καταρχήν τι σημαίνει πλεονάζουσα χωρητικότητα ή υπεραλίευση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στοχευμένα. Τα, οι δημόσιες ε, δαπάνες δεν έχουν γίνει με κανονικό τρόπο ε, και θα πρέπει να δούμε που τοποθούνται ακριβώς τις δυσκολίες και όταν λέτε ότι δεν έχουμε επαρκή δεδομένα ε, δεν έχουν υποβληθεί εκθέσεις, δεν έχουν τηρηθεί κανονισμοί ε, και ειδικά σε σχέση με τον κανονισμό για τα καύσιμα το τονίσατε, θεωρώ ότι είναι καλό να το ξέρουμε γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ε, θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό, ώστε να επιβάλλουμε τις αντίστοιχες κυρώσεις, να θεσπίσουμε αντίστοιχες κυρώσεις ή να αναπτύξουμε κάποια άλλα εργαλεία, ώστε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτές τις αθέμητες ε, πρακτικές. Γιατί εδώ στο Κοινοβούλιο δεν ε, ε, φτάνει το να κάνουμε τις σωστές σκέψεις. Θα πρέπει και οι χώρες μέλη να μας συνδράμουν και να εκπληρώνουμε σωστά τους στόχους. Τώρα, ένα ερώτημα. Σκέφτομαι όταν μιλάμε για, την, για τον παραπλησμό των σκαφών, θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε διάφορες μορφές αλίας, διαφόρων τύπων αλλιευτικά σκάφη, ε, διάφορες αλλιευτικές δυνατότητες και διάφορους τρόπους αλλιεύσης. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εφόσον έχει αποδειχθεί σε μια χώρα μέλος ότι ε, έχουν εξεταστεί όλα αυτά τα πράγματα και έχει διαπιστωθεί ότι έχει μειωθεί η υπεραλίευση, η πλεονάζουσα χωρητικότητα, δηλαδή υπάρχουν τόσα αλευτικά σκάφη ούτως ώστε ε, να γίνεται η αλήψη κατά τρόπο που να μπορούν να επιβιώσουν κανονικά, να ζήσουν κανονικά οι αλείς, να έχουν επαρκείς πόρους, ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της εισαγωγής νέων μηχανών στα αλληλευτικά σκάφη. Είπατε ότι έχει υπάρξει μια μείωση των θέσεων απασχόλησης 70.000. Ε, ε, είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια και ε, νομίζω ότι σε σχέση με τα μελλοντικά εργαλεία που θα εφαρμόσουμε θα αυξηθούν, θα μειωθούν μάλλον ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Ε, ξέρετε πώς θα μπορούσαν να αντιστανιστούν αυτές οι απώλειες από κοινωνικές άποψεις. Ποια ταμεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν όσους πλήττονται από αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, υπάρχει μια υγιής αλία, όπως λέγεται, αλλά ίσως ε, θα μπορούσε να ενδεχομένως εμφανίζει για ένα μεταβατικό διάστημα κάποια οικονομικά προβλήματα αλλά ενδεχομένως αργότερα να οδηγήσει σε καλά οικονομικά αποτελέσματα. Για, αυτά τα, για αυτό το μεταβατικό διάστημα ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να προτείνουμε κάποιες ενισχύσεις, κάποιες βοήθειες. Ε, μπορείτε να εξετάσετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις ή μονάδες να δοθούν κάποιες βοήθειες κατά τη μεταβατική περίοδο. Λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι είμαι ευγνώμων για αυτή την έκθεση γιατί νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε μελλοντικά κάποια από τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρόντουστ. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ επίσης τον κύριο Λαζάρου η Γερμανία δεν είναι μια μεγάλη ελευτική χώρα ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζουμε την εξής κατάσταση. Όσον αφορά τα ΤΑΚ, ή τις ε, αλληλευτικές μας ε, επιχειρήσεις έχει υπάρξει μια ισορροπία και χαίρομαι που η σχετική σταθερότητα στις βόρειες ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα τάκ, δηλαδή τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα και την κατανομή στις διάφορες ε, χώρες μέλη θα συνεχίσει να ισχύει αυτό το σύστημα γιατί με τον τρόπο αυτό κάπως κατευνάζεται όλη η κατάσταση σε όλες τις χώρες μέλη κατευνάζονται οι ανησυχίες. Και μιλήσαμε για την ε, ζώνη των, ε, των 12 μιλίων ε, και για τη συμφωνία που υπάρχει με τους αλείς, ούτως ώστε να μπορούν να αλλιεύουν μπροστά στις ακτές των διαφόρων χωρών μελών. Τώρα, υπάρχει το θέμα των μεταβιβάσιμων ε, δικαιωμάτων, τα οποία όμως ε, ορίζονται επακριβώς σε σχέση με συγκεκριμένα ληφτικά σκάφη, όχι με επιχειρήσεις ή με άτομα. Και πραγματικά εδώ φτάνουμε στο κεντρικό θέμα το οποίο συζητούμε εδώ και στο οποίο αναφέρθηκαν και ο κύριος Καντέκ, ε, ο κύριος Στίβενσον, όλοι όσοι μίλησαν προηγουμένως. Χρειαζόμαστε μια ε, ακριβή ανάλυση σχέση με την λευτική ικανότητα, δηλαδή ε, πώς, τι θα κάνουμε με το ληφτικό μας στόλο στην Ευρώπη. Αυτό είναι το α και το ω όταν μιλούμε για ποσοστώσεις και λέμε ποιες ποσότητες θα πρέπει να έχει το κάθε μέλος ε, και ποια θα πρέπει να είναι η ελευτική ικανότητα του κάθε στόλου. Ε, και το θέμα της υποδύναμης των μηχανών είναι καθοριστικό. Ε, με τις μηχανές που έχουμε σήμερα μπορούμε να λεύουμε και στην τα είδη αλλά θα πρέπει να αναφέρεται το όριο της υποδύναμης κινητήρα. Και ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε πραγματικά ε, ξεκάθαρα, ξεκάθαρες δηλώσεις. Δηλαδή, πρώτον, χρειαζόμαστε ποσόστοση, ε, άδειε δικαιώματα επίσης, αλλά θέλουμε επίσης ξεκάθαρα, ξεκάθαρες διατάξεις για το πόσο θα πρέπει να είναι η υποδύναμη των κινητήρων, το μάτι των ε, δικτυών κλπ. Ε, η εποπτεία της αλίας είναι το α και το ω εδώ. Και έτσι όπως έχουμε καθορίσει τους κανόνες, ε, είναι ένα τεράστιο σύστημα κανόνων και όταν κανείς βγει στην ανοιχτή θάλασσα, όταν ε, χρειάζεται να πάει να πεφθεί σε διάφορες υπηρεσίες. Ε, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, το πώς θα πρέπει να ζυγιστούν τα ψάρια επί του σκάφους κλπ. Η, ε, ε είναι ξεκάθαρη είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή και το πώς διενεργούνται οι έλεγχοι όσον αφορά τη ζώνη των τριών μιλίων, για παράδειγμα. Ε, και υπάρχουν και διάφορες αρμόδιες ε, αρχές. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, διάφορες δυνατότητες να εφαρμοστούν όλα αυτά. Δηλαδή, η έκθεση είναι σημαντική, αλλά θα ήθελα να πω ε, ξεκάθαρα ότι τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα αλίες, δηλαδή δικαιώματα αλίες τα οποία μπορούν να πολλούνται, δεν είναι υπέρ του συμφέροντος της Γερμανίας από τη μία, αλλά και της ε, παράκτιας αλίες μικρής κλίμακας. Γιατί θα είχαμε μια, στην περίπτωση αυτή πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση και όλα θα είναι συνάρτηση του κέρδους. Γιατί το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, παράκτη αλία μικρή κλίμακα που να έχει έναν αυθεντικό χαρακτήρα και εδώ ο τουρισμός παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο. Και ε, αυτά σε διαφορετικά αδύναμες ε, περιοχές όπου υπάρχει αυτή η αλία μικρής κλίμακας, αυτά είναι τα ζητήματα που, τίθενται γιατί υπάρχει η σύζευξη αλίας και τουρισμού. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Άρα λοιπόν όσον αφορά τα μεταβάσιμα δικαιώματα εγώ είμαι ε, ξεκάθαρα κατά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, διατάξεις, κάποιοι κανόνες που να μπορούν να επιτρέπουν μια δυνατότητα ε, βιωσιμότητα στα μικρές επιχειρήσεις. θα πρέπει οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν την αλία όταν συνταξιοδοτηθούν οι πατεράδες τους. Επίσης να υπάρξουν κάποια δυνατότητα στο τουριστικό τομέα. Να, για παράδειγμα να κάνει κανείς ε, διακοπές ε, πάνω σε ένα ε, αλευτικό σκάφος για παράδειγμα ή σε μια περιοχή όπου υπάρχει αλία. Υπάρχουν τις δυνατότητες. Και θα ήταν πολύ καλό να υπάρξει και μια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με όλα αυτά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ερνέστο Πένιας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να αποφανθεί στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού γιατί και η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως την ανάλυση του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί αυτή η έκθεση δίνει την έμφαση σε ορισμένα προφανή σημεία που χαρακτηρίζουν την ε, αλληλευτική πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας και αυτή η έκθεση μας κινητοποιεί ώστε να ακολουθήσουμε το στόχο μεταρρύθμισης της παρούσας πολιτικής. Είναι προφανές ότι κατανοούμε ότι η υπεραλίευση συνεχίζει να παραμένει θεμελιώδες πρόβλημα για την ε, αλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υπεραλίευση μας εμποδίζει ακριβώς να διατηρήσουμε τα βιολογικά υποθέματα σε ένα ε, βιώσιμο επίπεδο καθώς και να διατηρήσουμε τα έσοδα των αλλαίων είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Αλλά όποια και αν είναι η δυνατότητά μα να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα τη υπεραλίευση και όποια και είναι η εμβέλεια τη τη χωρητικότητα, δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι το φαινόμενο αυτό υπάρχει. Και εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα τη εκμετάλλευση των πόρων και η μια αποδοτικότητα του Ευρωπαϊκού Στόλου είναι μια έμεση ξεκάθαρη απόδειξη αυτού του γεγονότος, καθώς και το γεγονός ότι πολλοί από εσά ε, συνεχίζετε να ζητάτε ε, μια βοήθεια όσον αφορά την απόσυρση των αληθικών σκοφών και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα κάποιο επίπεδο υπεραλίευσης, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν αναγκαία η απόσυρση των αληθικών σκαφών. Καταλαβαίνουμε ότι η απόσυρση των ληφτικών σκαφών είχε ήδη κάποιες θετικέ επιπτώσεις αλλά δεν, και δεν αφιβάλλουμε ότι σε πολλέ περιπτώσει υπήρξε θετική αυτή η διαδικασία. Αλλά αναφίβολα αυτό το οποίο είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να αναλύσουμε την αξία αυτού του εργαλείου και να δούμε κατά πόσο η δαπάνη των 2.700.000 ε, συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυση του προβλήματος. Στην ανάλυση μας συμπίπτουμε με την ανάλυση του ελεγκτικού συνεδρίου, δηλαδή με όρους ε, κόστους και ωφέλες, το να δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα για την απόσυρση χωρίς να επιλύεται το πρόβλημα δεν είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή και ε, στη βάση αυτή προτείναμε την, ε, ε, την ε, πάυση της επιδότησης, της ενίσχυσης των, για την απόσυρση των σκαφών. όποια, είναι ο ορισμός που δίνουμε στην υπεραλήψη, είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε ένα ορισμό που να λαμβάνει υπόψη τι τεχνικέ εξελίξει. Και εδώ συμπίπτουμε με την ανάλυση του ελεκτικού συνεδρίου ότι πέρα από την ονομαστική μείωση της ε, πλεονάρωσης χωρητικότητας της υπεραλίευσης που έγινε τις προηγούμενες ε, δεκαετίες είναι πιθανόν ότι αυτή η ονομαστική μείωση αντισταθμίθηκε εν μέρη ή πλήρως από την βελτίωση της τεχνολογίας τελευταία σκάφη. Δηλαδή με όρους κόστους ωφέλειας και σε σχέση με τις ε, δημόσιες δαπάνες κατασπαταλήσαμε, ε, διασπαθήσαμε τους δημόσιους πόρους και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει επιληθεί, ε, και το θέμα είναι δεν έχει επιληθεί ακόμα το πρόβλημα της τη χωρητικότητας. Λοιπόν, η Επιτροπή προσπαθεί λοιπόν με αυτή την εφετηρία να επιλύσει ορισμένα από τα θέματα που αναφέρει και έκθεση η δυσκολία μέτρησης, η δυσκολία υποβολής αιτήσια έκθεσης εκ των χωρών μελών εν σχέση με τη δική του αλληλευτική ικανότητα και σε συνάρτηση με τα διάφορα μέτρα. Ε, έχουμε θεσπίσει κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές εν σχέση με την ε, υποβολή εκθέσεων για την αλληλευτική ικανότητα της κάθε χώρας μέλους κλπ. Και βεβαίως ε, όλοι μίλησαν για την ανάγκη ενός καλύτερου ορισμού της πλεονάς χωρητικότητας ή υπεραλίευσης. Και θα προσπαθήσουμε να σας προτείνουμε κάποιον πιο κατάλληλο ορισμό. Λοιπόν, ε, στη βάση αυτής της ανάλυσης ε, προτείνουμε ως λύση τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα, θέμα για το οποίο μιλήσατε εσείς. Η Επιτροπή κατανοεί ότι παρόλο που δεν ε, εμφανίζουμε το σύστημα αυτών των μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων σαν πανάκια, ε, θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει με ένα πραγματικό ρεαλιστικό τρόπο σε ορισμένε χώρε. Και εκεί όπου έχει εφαρμοστεί, γενικά, σε γενικέ γραμμέ, τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά και μπόρεσε να υπάρξει μια θετική προσέγγιση του ζητήματος της υπεραλίευσης και αυτό χωρίς διασπάθηση των δημόσιων πόρων. Κάτι που έχει μεγάλη σημασία για μας. Λοιπόν, η Επιτροπή δεν προτείνει βεβαίως ε, την προσέγγιση one size fits all, αλλά θεωρεί ότι τα μεταβιβάσιμα, το σύστημα μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων ε, μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα στην πραγματικότητα της κάθε χώρας μέλους. Και αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής. Βεβαίως, και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και πολλοί από εσά αναφερθήκατε στο ζήτημα της διαφορετικής βοήθειας, η Επιτροπή κατανοεί ότι όποια και είναι η μείωση της ε, πλεονάσεως χωρητικότητας που θα υπάρξει στο μέλλον, υπάρχει ένα πρόβλημα ε, απώλειας των θέσεων απασχόλησης που θα πρέπει να αντισταθμιστεί με κάποια μέτρα του Ταμείου Αλίας. Ε, και ε, η Επιτροπή στην πρόταση κανονισμού όσον αφορά το Ταμείο Αλίας ε, βάζει την έμφαση ειδικά όχι στον παροπλισμό που όπως όλοι γνωρίζουμε ε, μειώνει τον ελευθερικό στόλο, αλλά δίνει έμφαση στην προαγωγή συμπληρωματικών οικονομικών δραστηριοτήτων ή εναλλακτικών προς την αλληλεία ούτως ώστε να προαχθεί ενεργά η απασχόληση στις ζώνες όπου μειώνονται οι ελευτικές δραστηριότητες. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στι ορισμένε παρεμβάσει των βουλευτών, συγκεκριμένα σε ένα θέμα που ανέφερε ο κ. Στίβενσον, που για την Επιτροπή είναι μέγιστη σημασία και είναι η αναφορά που έκανε και που συμμεριζόμαστε πλήρω στο πρόβλημα της ε, μέτρησης της υποδύναμης των ελευθερικών σκαφών. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι έχει δίκιο η κυρία ε, Δαμανάκη την προηγούμενη, είχε δίκιο η κυρία Δαμανάκη την περασμένη Δευτέρα όταν είπε ότι ό,τι κι αν ε, σκεφτούμε για τη δυνατότητα εισαγωγή κάποιων ε, βοηθειών, ενσύσεων για την απόσυρση των σκαφών, θα πρέπει οι χώρες μέλη να έχουν τη δυνατότητα να καταμετρούν και να ελέγχουν επαρκώς την υποδύναμη των κινητήρων των αλληλευτικών σκαφών γιατί αυτές, ε, αυτά τα χρήματα για τον εξοπλισμό των σκαφών ε, χορηγούνται χωρίς ακριβώς ε, να υπάρχει προϋπόθεση της, του ελέγχου της ε, μηχανής των αληφτικών σκαφών. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ε, ενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων προκειμένου να χορηγούνται αυτές οι βοήθειες για τον εξυγχρονισμό. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρένιας. Μετά από τόσες ε, παρεμβάσεις κύριε Λαζάρου να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους τους παρεμβαίνοντες για τις παρατηρήσεις τους και τις ερωτήσεις. Πραγματικά είναι συναρπαστικές. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να απαντήσω. Βεβαίως, οι περισσότερες είναι περισσότερο πολιτικής φύσεως παρά τεχνοκρατικής. Κάτι που δεν είναι ακριβώς ε, το πεδίο αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνέδριο έχει προσπαθήσει στην ειδική έκθεσή του να παρουσιάσει γεγονότα βασισμένο στα πορίσματα των ελέγχων και θα έχετε παρατηρήσει ότι στην έκθεση δεν κάνουμε συνολικές συστάσεις. Στόχος μας, όπως σε κάθε ειδική έκθεση, είναι πριν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ε, νομοθετικές αρχές να δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να συζητηθεί το υλικό που διαθέτουμε. Να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις δηλαδή σε οποιοδήποτε ζήτημα, όχι μόνο στην Αλία. Σε αυτή την περίπτωση επικρίνουμε, ναι, επικρίνουμε την ε, κοινή ελευθερική πολιτική σε αυτά τα μέτρα όπως λειτουργεί, αλλά έχουμε πετύχει το δικό μας στόχο. Κάτι που είναι σε κάθε περίπτωση στόχος μας. Να εξυπηρετήσουμε τις συζητήσεις, τις διαβουλεύσεις, ώστε να ληφθούν και κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις και από εσάς. Και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορεί να συσχετίζονται με την κοινή, κοινή αλληλευτική πολιτική. Βεβαίως είναι σημαντικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες. Βεβαίως και αποτελεί μέρημνα όλων. Οι Ευρωπαίοι να έχουν δουλειέ, ιδίω σε τόσο δύσκολους καιρούς. Ανέφερα μάλιστα συγκεκριμένα και τη μείωση των θέσεων εργασίας. Τώρα, μετά από αυτή την εισαγωγή θέλω να προχωρήσω λέγοντας ότι η κυρία Ρόντουστ την ε, δική της παρέμβαση στα εισαγωγικά της σχόλια εξήγησε το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου από μια διαφορετική σκοπιά, μπορεί και καλύτερη από εμένα τον ίδιο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν λέμε παροπλίστε και αποσύρτε. Όχι, λέμε καλύτερη στοχοθεσία. Ο τρόπος που έχει εφαρμοστεί το μέτρο αυτό τώρα δεν έχει δώσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Αυτά που προσδοκούσαμε. Το να μιλάμε για το θέμα της δυνατότητας, της πλεονάζουσας δυνατότητας. Καθοριστική έννοια στην ε, ισχύουσα κοινή λευτική πολιτική. Δεν είναι κάτι που δεν, δεν πρέπει να υπάρχει, να το ξανασκεφτούμε όμως, αυτό λέμε. Να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας, διότι αν οι πολιτικές βασίζονται σε τέτοιες έννοιες όπως οι δυνατότητες, οι πλεονάζουσες δυνατότητες, Καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει διαφορετική διαφορά 200.000 τόνους στη χωρητικότητα σε σχέση με αυτό που εννοούσαμε αρχικά, πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Δεν λέμε να μεταρρυθμίσουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική αποκλείοντα την έννοια τη πλεονάζουσα δυνατότητα. Τώρα, τα Τα σημεία που, στα, στα οποία στάθηκαν οι βουλευτέ, να ξεκινήσω από τον κύριο Κάντεκ, η υπερβολική δυνατότητα, η πλενόσα δυνατότητα και η υπερχωρητικότητα είναι καθοριστική σημασία στη σημερινή κοινή αλληλευτική πολιτική. Με ρωτήσατε ποιο είναι ο ορισμό. Είναι η δυνατότητα του αλληλευτικού στόλου να αλλιεύει πέραν όμως του ποσού, του, της ποσότητας, που βάσει επιστημονικών ε, στοιχείων, τι δεν είναι αυτό. Είναι Αλλά εφόσον, αλλά μπορεί, η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά το σύνολο των αλλιευτικών ευκαιριών. Αυτό είναι η πλεονάζουσα δυνατότητα. Όμως, ό,τι αφορά την, την απόσυρση και τον παροπλισμό, δεν είπαμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο αυτό. Απλώς λέγαμε να υπάρξει καλύτερη στοχοθεσία. Υπάρχουν παραδείγματα στην έκθεση που φανερώνουν ότι δεν υπήρξε στόχη, σωστή στοχοθεσία. Σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό, Συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει να εξυγχρονιστούν τα ελληνικά σκάφη, αλλά μέσω στη στόχοθεσία, ε, όπως ήταν ο αρχικός στόχος για την αύξηση του επίπεδου ασφάλειας, για τα ζητήματα τα υγειονομικά. Όμω, κάποια από τα προγράμματα εξυγχρονισμού αυτού τελικά αύξησαν και τη χωρητικότητα των σκαφών, τη δυνατότητα αλίευση των σκαφών. Πάλι έχουμε θέμα στοχοθεσία. Στην έκθεση αυτή δεν τοποθετούμαστε ως προς το θέμα των μεταβιβάσιμων ε, αλληλευτικών δικαιωμάτων. Δεν λέμε αν θα πρέπει ή όχι να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Το μόνο που λέμε είναι ότι υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα και πρέπει να τα αποσαφηνίσουμε. Αντιφατικά στοιχεία σε σχέση με την υπάρχοντα, τον ισχύοντα κανονισμό της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και διαβάζω αυτό που σας είπα και στην παρουσίασή μου. Η κοινή αλληλευτική πολιτική δίνει αντιφατικά μηνύματα για το θέμα αυτό. Ε, ο κανονισμός, ο βασικός κανονισμός του, ε, του Συμβουλίου του 2002 προβλέπει συγκεκριμένε δυνατότητε για τα λιευτικά σκάφη, όμω άλλο κανονισμό επιτρέπει την επανακατανομή των ποσοστώσεων. Πρέπει λοιπόν να αποφασιστεί τι από τα δύο θα ισχύσει. Και βάσει των ε, πορισμάτων του ελέγχου μας, το αναφέρει και η έκθεσή μας, σε δύο τουλάχιστον χώρες αναφέρεται ότι το πρόγραμμα των μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων εφαρμόστηκε και έτσι εξισορρόπησαν μπόρεσαν να εξισορροπήσουν τι αλληλευτικέ δυνατότητε με τις υπάρχουσες αλληλευτικέ ευκαιρίε. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις αυτό. Όμω, λογικό είναι οι ελεγκτές που είναι εδώ για να σας συνδράμουν, να σας διευκολύνουν στις διαβουλεύσεις σα, να σας διαθέσουν και όλες τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μα. Προχωρώ στις ερωτήσεις του κυρίου Στίβενσον. ελέγχθη ότι υπάρχει 30% αύξηση στα εμπορεύσιμα αλληλευτικά αποθέματα βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών. Τεχνικότατη ερώτηση και η απάντησή μου είναι ότι βασιζόμενοι στις στα στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής από το 2009, ότι το 90% των ειδών είναι αντικείμενο υπεραλίευσης και το 30% είναι κάτω των βιώσιμων ε, επιπέδων, βιώσιμων ποσοστών και μάλιστα μέσω των πληροφοριών της ειδική μας έκθεσης, στατιστικά στοιχεία που έχουμε από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών. Αυτά ήταν τα στοιχεία που διαθέταμε εμεί. Δεν ξέρω εσεί από πού αντιλήσατε την πληροφορία σα, δεν μπορώ να την αμφισβητήσω. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω περαιτέρω. Εάν σωστά το σημείωσα, μιλήσατε για τις ενισχυμένες μηχανές, για τις επί του σκάφους επενδύσεις. Αυτό εμείς δεν το αναφέρουμε στην έκθεσή μας. Εμέσως, πιστεύουμε όμως ότι τέτοιου είδους επενδύσεις, οι ανπλού επενδύσεις, μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αύξηση της δυνατότητας υπεραλίευσης. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που έχουν οι κλιματικές αλλαγές στα αλληλευτικά αποθέματα, αυτό δεν το καλύψαμε στο πεδίο του ελέγχου μας. Δεν θα το σχολιάσω λοιπόν. Αλλά αφήνοντας κατά μέρος την ιδιότητα που έχω σε πιστεύω ότι σίγουρα οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν επηρεάσει όλες τους ζώντες οργανισμούς, όπως έχει συμβεί με τα ψάρια και με τα δάση υποθέτω. Δεν ξέρουμε τώρα σε τι βαθμό. Χρειάζονται περαιτέρω επιστημονικές μελέτες από αυτού. Να περάσω στα ερωτήματα του κυρίου Γκάλαχερ. Η Ιρλανδία δεν επελέγει. Όπως προανέφερα, στόχος ήταν να μελετήσουμε τα κράτη-μέλη που συνολικά κατέληγαν στις μεγαλύτερες τιμές στον από απόψη προπολογισμού ποσών. Εκείνη τη στιγμή δεν μελετούσαμε την, τον παροπλισμό, αλλά το ε, συνολικό ποσό. Τα συνολικά ποσά δηλαδή. Και πάλι, το θέμα των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών δικαιωμάτων, Κατάλαβα την παρατήρησή σας, όπως και κάποιοι άλλοι σας συνάδελφοι, το είπατε κι εσείς, αλλά εμείς δεν τα προωθούμε τα μεταβεβάσιμα αλληλευτικά δικαιώματα. Δεν είμαστε υπέρ, υπέρ τους. Αλλά νομίζω τα καταλαβαίνετε καλύτερα και από μένα. Υπάρχουν υπέρ και κατά σε σχέση με τα αλληλευτικά δικαιώματα. Πρέπει απλώς να αποσαφινιστούν στους κανονισμούς. Και έχουμε και την περίπτωση των συγκεκριμένων δύο κρατών μελών. Κύριε Γκάλαχερ, δίκιο έχετε. Σε ό,τι αφορά τον παροπλισμό των σκαφών και τα μεταβιβάσιμα αλληλευτικά δικαιώματα, δεν τοποθετούμαστε εμείς στην εκθεσή Δεν λέμε να εγκαταλειφθούν τα προγράμματα παροπλισμού ή όχι, απλώς να ε, σχεδιαστούν και να οργανωθούν καλύτερα. Τώρα, οι ερωτήσεις της κυρίας Ρόντουστ. Εάν σωστά τα σημείωσα, ρωτήσατε, εάν έχουμε τελικά στα χέρια μας αποδεικτικά στοιχεία από οποιοδήποτε κράτος μέλος, ότι ο παροπλισμός, τα προγράμματα μάλλον παροπλισμού, συνέβαλαν στην εξισορρόπηση των αλλιευτικών δυνατοτήτων με τις αλλιευτικές ευκαιρίες. Αυτό ρωτήσατε. Εξ όσων γνωρίζω, αλλά μπορεί και να ασφάλω, όχι, δεν ε, είχαμε τέτοια στοιχεία από κανένα κράτος μέλος. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει σε αρκετά είναι οι βοήθειες που καταβλήθηκαν για τον παροπλισμό να μην συνοδεύονται από εκπλήρωση των ε, προϋποθέσεων. Για το κατά πόσον γνωρίζουμε τι μεταρρυθμίσεις καλό θα ήταν να προταθούν στα πλαίσια της γενικότερης προτινόμενης μεταρρύθμισης, θα σας παραπέμψω στην εισαγωγή. δεν είναι δική μας ε, αρμοδιότητα, ούτε δικό μας προνόμιο να κάνουμε τέτοιου είδους συστάσεις. Εσείς θα πρέπει να το κάνετε. Να συνεχίσω. Σε ό,τι αφορά τη δική σας την παρατήρηση για το κατά πόσον θα έπρεπε να υπάρξει σε μεταβατική περίοδο οικονομική στήριξη εφόσον το πρόγραμμα μεταβιβάσιμων ληφτικών δικαιωμάτων τελικώς εφαρμοστεί και πάλι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Εάν οι υπεύθυνοι για την νομοθεσία κατά τις διαβουλεύσεις τους αποφασίσουν ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα τελικά θα πρέπει να υλοποιηθεί, τότε εκείνοι θα πρέπει και να αποφασίσουν ποια είναι η βέλτιστη μέθοδος εφαρμογής του. Να προχωρήσω τώρα στις δηλώσεις του κ. Καν για τα μεταβιβάσιμα αλληλευτικά δικαιώματα. Νομίζω Με τις απαντήσεις που έδωσα για τα προηγούμενα ερωτήματα σας έχω ήδη απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν uh, θέλει να, δεν η κυρία Ρόντουστ. Όπως είπατε και εσείς κύριε Λαζάρου ήταν ε, δύσκολες οι ερωτήσεις, ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. γνωρίζαμε ότι ήταν ε, επικριτική η έκθεσή σας είχε λοιπόν σημαντικό ενδιαφέρον για μας να προσέρθετε εδώ και να συζητήσουμε μαζί σας και για τα μέλη μας που ήταν παρόντα νομίζω ότι τα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο συγκεκριτής μας κύριος Μιλάνα θα υποβάλει σχέδιο γνωμοδοτήσεως για το θέμα αυτό τον Μάιο. Στο μεταξύ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι που προσήλθατε και εδώ λύγει το θέμα αυτό της τη διαταξής μας. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης γιατί είχαμε αναβάλει το 15, 16 και 17 και επομένως ερχόμαστε στο 18 έκθεση δηλαδή σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αλίας στην Βρετάνη από τις 20 Φεβρουαρίου έως 22 και μου λένε ότι τέσσερα μέλη δεν μπορούσα να διαβάσω καλά, νόμιζα ήταν εννέα στην αρχή αυτό. Τέσσερα λοιπόν μέλη συμμετέσχων με τα από πρόσκληση του Αλάν Καντέκ του στον οποίο θα δώσω το λόγο για να προχωρήσει αμέσως να μας εξηγήσει τι έγινε στην επίσκεψη στη Βρετάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τόσοι βουλευτέ ήταν μαζί μα στη Βρετάνη, όσοι είναι και εδώ στην αίθουσα. Ε, Ένα, δύο, τρει, τέσσερι για να μετρήσω. Πέντε, ε, λίγο παραπάνω. Απλώ για να σα πω ότι όσοι δεν ήρθαν, έχασαν. Το ίδιο το ταξίδι πήγε πολύ καλά. Πρώτα την πρώτη μέρα. Παραστήκαμε στην αλίευση πελερινίτσας, σαν ζάκι όπως λέγονται στα γαλλικά, στην, στον κόλπο του Σάμπριε, με δίχτυα, όχι με βιομηχανικό σκάφος, ε, παραδοσιακή αλία και υπόδειγμα τη σωστή διαχείριση ενό τέτοιου αποθέματο. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα επέτρεψε να. Θα μας επιτρέψει μάλλον να συνεχίσουμε χωρί να κάνει πηγαδάκια. Έτσι, Ερνέστο. Ερνέστο. Και πάλι ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας επιτρέψει να συνεχίσουμε. Κύριε Πένιας, θα παρακαλούσα τον Ερνέστο να σοπάσει. Ερνέστο, σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Συνεχίζω λοιπόν. Να σας πω ότι μετά πήγαμε στην Πρέστ μας παρουσιάστηκε εκεί η μεγαλύτερη ένωση παραγωγών της Ευρώπης. Οι αλλοί της Βρετάνης με 800 σκάφη μας εξήγησαν πώς έχουν οργανωθεί και έπειτα ήμασταν καλεσμένοι στην Ιφρεμέρ. Στο νευραλγικό σημείο αυτό, κάποια χιλιόμετρα από την Πρέστ, εκεί συναντήσαμε ε, επιστήμονες που μας παρουσίασαν και τις ανησυχίες και τις ελπίδες τους για το μέλλον της Αλίας. Μας παρουσίασαν και οι μεν και οι δε τις δικές τους απόψεις για την ανάγκη μεταρρύθμισης της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, αλλά με τρόπο ευφύ και σκόπιμο. Λαμβάνοντα υπόψη και τι επιστημονικέ απόψει που εκείνοι μα παρουσιάζουν και τι απόψει των αλλιών. Έπειτα επισκεφτήκαμε την Οκεανόπολη. Αξιοθέατο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ε, κάποιοι από εμά ανακάλυψαν, αν εγώ τα γνώριζα βέβαια ήδη, ένα χώρο που είναι αφιερωμένο στη θάλασσα, ιδίως στην Αλία, μας ε, υπεδέχθη ο υπεύθυνο, ε, ο αξιωματικός, αξιωματικός μάλλον στην ιδιωτική του κατοικία, ε, και την επόμενη μέρα εγώ και άλλοι συνάδελφοι, ο κ. Μιλάνα, και άλλοι είχαμε συνάντηση με ενώσει αλλιέων, συναντήσεις μάλλον με ένωση αλλιέων και συζητήσαμε με τους ίδιους τους αλλιείς για το γεγονός ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη τη μεταρρύθμιση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής τη ζωή των αλλιών, την καθημερινότητά του και θα πρέπει να είναι υπέρ τους, αλλά και σε καμία περίπτωση εναντίον τους, όπως και εγώ υποστηρίζω διαρκώς. Και μετά χωριστήκαμε. Χωριστήκαμε για να γυρίσουμε ο καθένα σπίτι του. Σας διαβεβαιώ ότι κάθε φορά μεταξύ αυτών των συναντήσεων και πολύ καλά γευματίσαμε και διπνήσαμε με πολύ καλή ατμόσφαιρα και μάθαμε και πολλά. Σας βεβαιώνω λοιπόν το ταξίδι μας και επικοδομητικό ήταν και πολύ αποδοτικό από την άποψη του φαγητού. Σας ευχαριστούμε κύριε Καντέκ. Πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη. Uh, ε, Λυπούμε που δεν μπόρεσα να συμμετάσχω, αλλά έχω πάει πολλές φορές στη Βρετάνη. Δεν ξέρω αν κανείς επιθυμεί να σχολιάσει για αυτό το σημείο. ή αν όχι, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 19, διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα από δική μου, από μου πλευράς, δεν ξέρω, ούτε από δική σας. Άρα πάμε στο σημείο υπερθμό 40, οι αποφάσεις των συντονιστών που έχουν διανεμηθεί σε όλους και υποθέτω ότι υπάρχει συμφωνία. Άρα πάμε στο σημείο 21, την προσεχή συνεδρίαση που είναι στις 23 και 24 Απριλίου. Περιμένουμε ε, να σας δούμε εκεί. Μία ερώτηση. 23 είναι Δευτέρα απόγευμα. Δεν ξέρω, θα λάβει χώρα, θα, γίνει, θα διεξαχθεί ψηφοφορία τη Δευτέρα, ε, τη Δευτέρα απόγευμα ή θα γίνει την Τρίτη. Απάντηση, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ψηφοφορία την Τρίτη γιατί βολεύει περισσότερο τα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε όλους.